οι αρμόδιες επιτροπές υπέβαλαν ε, διορθωτικά για έξι κείμενα σύμφωνα με τον κανόνα 231 παραγραφός 4. σε περίπτωση λοιπόν που ε, αυτό υποβάλλεται από 40 τουλάχιστον βουλευτούς τα πρακτικά και τα κείμενα αυτά θα τα βρίσκεται στις σχετικές ε, σελίδες που δημοσιεύονται στο διαδικτύο για την Ολομέλεια. Εγκρίνονται λοιπόν και οι τίτλοι των ε, νομοθετικών αυτών πράξεων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα για την Ολομέλεια. Και τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, στο σχέδιο εργασίας.